Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά της συνεδρίας αυτής θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρία του Κοινοβουλίου και τα ψηφίσματα αυτά θα